Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, δέκα ημέρες μετά τον τυφώνα Χαϊάν που σάρωσε με πάνω από 300 χιλιόμετρα ολόκληρες εκτάσεις της Φιλιππίνης για εκατοντάδες χιλιάδες επιζώντες παραμένει δραματική η κατάσταση. Γνωρίζετε όλοι τις εικόνες ε, απελπισμένων ανθρώπων που δεν έχουν πόσιμο νερό, καθόλου φαγητό και είναι υποχρεωμένοι να διεκτερεύουν στην Ήπεθρο. Έχει αρχίσει να φτάνει η βοήθεια αλλά παραμένουν ορισμένες περιφέρειες αποκομμένες από τον έξω κόσμο είναι ε, περίγραπτο το χάος που επικρατεί εκεί. Ε, η ε, βοήθεια και τα συνεργεία διάσωσης αναζητούν αγνοωμένους, αγωνίζονται μέσα στα συντρίμια, άνθρωποι να επιβιώσουν και χρειάζεται βοήθεια διεθνής από το εξωτερικό. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να βοηθήσει τον κόσμο αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα που το έχει τεράστια ανάγκη και για την ανοικοδόμηση των χωριών και των πόλεων που έχουν καταστραφεί χρειάζεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει και επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και πιο μακροπρόθεσμη έχει δεσμευτεί αλλά νομίζω ότι μπορούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε περισσότερα είναι δραματική η κατάσταση 11 εκατομμύρια άνθρωποι στις Φιλιππίνες πλήττονται από τις συνέπειες αυτού του τρομακτικού τυφώνα. Είναι δραματικά τα αριθμητικά στοιχεία. 660.000 άνθρωποι είναι άστεγοι, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Και σύμφωνα με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό είναι ακόμα 22.000 οι αγνοούμενοι, ενώ ο αριθμός των νεκρών θα το διαβάσατε, είναι πάνω από 2.500. Οι ε, οργανώσεις βοηθείας μας λέγουν ωστόσο ότι τα ε, στοιχεία αυτά τα νούμερα θα αυξηθούν οπωσδήποτε. Θα ήθελα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απευθυνθώ στους πληγέντες και να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ε, ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση και σίγουρα Είμαι βέβαιος ότι ε, μοιράζετε κι εσείς μαζί μου τα αισθήματα της αλληλεγγύης με τις οικογένειες και τα θύματα. Και θα σας παρακαλούσα να τηρήσουμε ενός λεπτού ε, σιγή. Και σας παρακαλώ να γερθείτε από τις θέσεις σας. Herzlichen Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να καλωσορίζω 150 μαθητές και μαθήτριες από 33 ε, χώρες. Καλωσορίσατε στη Euroscola. Είναι μια διημερίδα από χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και την Ουκρανία στα πλαίσια της Euroscola Euronest και θα συζητήσουν θέματα που ε, ενδιαφέρουν την ανατολική γειτονία. Είναι καλό να βλέπει κανείς νέους να συμμετέχουν το δημοκρατικό γίγνεσθε. Και είναι μακρύς ε, ο, ο διάλογος από τη δημοκρατία μέχρι την ε, εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συζητήσεις που είχατε. Ήταν πάρα πολύ ζωντανές, ε, με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος συμμετείχατε εκεί και δεν υπολείπεται σε τίποτα η δική σας συνέλευση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σε εύχομαι καλή επιτυχία στη ζωή σας και τη σταδιοδρομία σας. Επαναλαμβάνεται η σύνοδος, η περίοδος σύνοδου που ε, διακόπη στις 24 του μηνός Οκτωβρίου. Ο Σάνφος Τίερ έχει μια ερώτηση, παρακαλώ gospodine predsjednie jutros je oko one hundred tisua ljudi prolo kroz ili su iz vukovarske bolnice do memorijalnog groblja najvee masovne grobnice u europi. Ε, έκαναν πορεία στο Βούκοβα ε, και ε, είναι 22 χρόνια μετά τη μάχη. Για πρώτη φορά από τότε που είναι μέλος η Κροατία έρχεται αυτή η επέτειος της μάχης του Βούκοβα. Γι' αυτό ήρθε και ένας αριθμός Κροατών πολιτών σήμερα στο ημικύκλιο επισκέπτες και θα ήθελα εξ ονόματός σας να τους χαιρετήσουμε, να τους καλωσορίσουμε και να αποτίσουμε το σεβασμό μας στους πεσόντες στη μάχη του Βούκοβα. Τώρα έχει έρθει η ώρα να ζούμε όλοι σε μια ενωμένη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στία για τα όσα μας είπατε και την υπόδειξη αυτή. Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 24 Οκτωβρίου διατίθενται. Έχετε στάσεις, αντιρρήσεις, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα συνοπτικά πρακτικά. Ερχόμαστε στις ανακοινώσεις. Οι αρμόδιες αρχές της ε, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας με ενημέρωσαν για την εκλογή της κυρίας Γκαμπριέλη Στάουνερ από τις 30 Οκτωβρίου και της κυρίας Μπράιερ από την 31 Οκτωβρίου 2013. Ε, η κυρία Στάουνερ αντικαθιστά την κυρία Βάις Γκέρμπερ, ενώ η κυρία Μπράιερ την κυρία ε, ε, Μπραντνερ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ε, για τις εκλογές στο μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα επίσης και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού του Κοινοβουλίου σημειώνουμε την εκλογή της κυρίας Στάουνερ και της κυρίας Μπράιερ με τις αντίστοιχες ημερομηνίε και τη λαμβάνουμε υπόψη. Καλωσορίζω ορίζω τις συναδέλφους και θυμίζω ότι και η κυρία Στάουνερ και η κυρία Μπράιερ σύμφωνα ε, με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού θα συμμετέχουν ε, με πλήρη δικαιώματα ε, στα όργανα του Κοινοβουλίου μέχρι να εγκριθεί ή να προσβληθεί εντολή τους και με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχουν δηλώσει ότι δεν ε, κατέχουν κανένα αξίωμα που είναι συμβίβαστο με ε, το αξίωμα του Ευρωβουλευτού. Οι αρμόδιες πολωνικές αργές ε, έχουν υποβάλει αίτημα για άρση ασυλίας του κυρίου και Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού διαβιβάζεται το αίτημα αυτό ε, στην Αρμόδια Νομική Επιτροπή ε, από ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Ελευθερία και Δημοκρατία έχουν υποβληθεί αιτήματα για ορισμούς σε επιτροπές. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις θεωρούνται αυτοί οι διορισμοί εγκεκριμένοι. Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε ένα διορθωτικό σε ένα κείμενο που εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του κανονισμού αν δεν διαφωνήσει η προπάλλη ένσταση μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται. Το κείμενο θα το βρείτε στο Seance on Direct και θα δημοσιευτεί και ο τίτλος στα πρακτικά της παρούς συνεδρίασης. Σύμφωνα με το άρθρο 74 ε, του κανονισμού μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω ε, τα κείμενα που εγκρίθηκαν, δέκα τον αριθμό ε, και στα σημερινά πρακτικά θα δημοσιευθούν οι επικεφαλίδες. Ερχόμαστε τώρα στην έγκριση της σημερινής διάταξης ή στην τροποποίησή της και στη διάταξη των εργασιών. Εγκρίθηκε στις 13.11 σύμφωνα με το άρθρο 137 το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης και έχει διανεμηθεί. Οι πράσινοι θα ζητήσουν δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της συμφωνίας TTIP. Πρόεδρε, ο κύριος Κονπεντήτ, και κάτι για τη διαδικασία ως προς την ψηφοφορία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δύο πράγματα. Ναι, δεν έχω φτάσει στην Τετάρτη ακόμα, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, αλλά ήθελα να σας το πω ότι το ζητήσαμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Κονβέντιντ, δεν είμαστε στην Τετάρτη.